Και επ' αυτού έχει το λόγο καταρχήν η Επίτροπος, η κυρία Μάλμιστερν. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε τρεις εβδομάδες που απομένουν μέχρι την ε, δέκατη υπουργική διάσκεψη στην Αϊρόμπη. Μέσα στα πλαίσια και της 20ης επαιτίου από τη λειτουργία της ε, Ντόχα. Η διάσκεψη αυτή ε, λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ΠΟΕ. Maybe I should wait a few minutes. No? Μετά την επιτυχία της τελευταίας διάσκεψης στο Μπαλί, και την εμπορική συμφωνία διευκολύσεων θεωρήσαμε ότι θα φτάσουμε σε μια εκτενή συμφωνία σε σχέση με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα. Δυστυχώς πολλές χώρες ε, δεν ήταν σε θέση ή δεν επιθυμούσαν να φτάσουμε σε ένα συμβασμό σε σχέση με τις επιδοτήσεις, τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στο Ναϊρόμπι θα πρέπει να, ε, να διευκολύνουμε το έργο του ΠΟΕ. Για να μην υπάρχουν φραγμοί θα πρέπει λοιπόν μέσα στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα να αποφασίσουμε για το τι θα κάνουμε. Τώρα εργαζόμαστε στη Γενέβη για να συμφωνήσουμε επί τριών ζητημάτων, επί τριών στόχων που αποτελούν μέρος της αξιοπιστίας μας. Καταρχήν, μια συμφωνία για να υπάρχει ένα πειθαρχημένο πλαίσιο αγροτικών εξαγωγών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ε, πολύπλευρη λύση. Μαζί με τη Βραζιλία και τον ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε μια επίσημη πρόταση για να δούμε το θέμα των επιδοτήσεων εξαγωγών σε γεωργικά προϊόντα. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση συζήτησης και ένα συμβιβασμό και έτσι βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των γεωργικών, των αγροτικών μεταρρυθμίσεων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να φτάσουμε σε μια κοινή αγροτική πρόταση με τη Βραζιλία. Εργαζόμαστε λοιπόν επί του θέματος στη Γενέβη. Δεύτερον, θα πρέπει να καλύψουμε τα πιο ευάλωτα και φτωχά μέλη του ΠΟΕ. Δηλαδή μιλάμε για θέματα επιδοτήσεων και την ε, εξάλληψη τελωνιακών δασμών καθώς και των κανόνων διαφάνειας στον ΠΟΕ. Εάν φτάσουμε σε συνένεση θα πρέπει να φτάσουμε και σε μια συμφωνία για το τι θα κάνουμε μετά την Υπουργική Διάσκεψη. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Ο ΠΟΕ θα πρέπει να συνεχίσει την, ε, τις εργασίες για μη επιλυμένα ζητήματα που μπορούν να επιληθούν μέσω διεθνών σχέσεων και πολύπλευρων προσεγγίσεων. Θα χρειαστούμε όμως νέες ιδέες, διότι οι παλές προσεγγίσεις δεν ήταν καλές. Οι αναδιόμενες χώρες λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Παράλληλα θα πρέπει η υπουργική διάσκεψη να ανοίξει τις πόρτες σε νέα ζητήματα για τα μέλη του ΠΟΕ, έτσι ώστε να διαπραγματεύονται ζητήματα μέσα σε μικρότερες ομάδες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία αν θέλουμε ο ΠΟΕ να αποτελέσει βασικό παράγοντα επίλυσης ζητημάτων. Η επερχόμενη λοιπόν υπουργική διάσκεψη είναι πολύ σημαντική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 Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Λάγκε, το συνεισηγητή, και να ευχαριστήσω και την Επίτροπο και την ομάδα, ομάδα της, η οποία πρόφησε αυτή την πολύπλευρη εργασία. Από πλευράς ΕΛΚ πάντα στοιχηματίσαμε υπέρ των πολυμερών σχέσεων και πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προωθήσουμε το ρόλο του ΠΟΕ. Πρόκειται για συμφωνίες διευκόλυνσης του εμπορίου για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης όλων των χωρών. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι όσο μεγαλύτερο εμπορικό άνοιγμα υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη θα υφίσταται. Αυτό το δείχνουν και οι μελέτες. Η Υπουργική Διάσκεψη στο Ναϊρόμπι, όπως είπε και η Επίτροπος, αποτελεί ένα σημείο, ένα κομβικό σημείο για να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειάζεται να δημιουργηθεί απασχόληση τώρα περισσότερο από ότι ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι οι πολυμερείς σχέσεις θα πρέπει να συνυπάρχουν με τις διμερείς συμφωνίες, τις ε, περιφερειακές και τις ε, πολυμερείς μέσα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου όπως το TTIP για παράδειγμα ή η συμφωνία με το Μερκοσούρ έχει μεγάλη, έχουν μεγάλη σημασία διεθνώς για να συμβαδίσουν και να συμπληρώσουν το γύρο της Ντόχα και τον ΠΟΕ σε τομείς όπου ε, πολλές φορές οι πολυμερείς σχέσεις δεν τα καταφέρνουν πάντα. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Λάγκε. Κύριε... κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, καταρχά να ευχαριστήσω τον συνεισήγητη κύριο Ζάλμπα. Και αναρωτιέμαι κάθε πόσο στο Ναερόμπι ε, έχει σβήσει το φω ε, για την ε, Νόχα. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι δεν θέλουν καν να μιλήσουν για το θέμα αυτό κάποιοι. Και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν βλέπω ο αναπτυξικό ε, γύρο τη Ντόχα και το γύρο του ΠΟΕ να μπορέσουμε να τον αναπτύξουμε περαιτέρω και να ε, καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα εργασία για πέρα από τον αερόμπιο, όπω είπε η Επίτροπο, αν δεν ε, αναφερθούμε θετικά και δεν βάλουμε ένα θετικό σημάδι σε αυτέ τι διαπραγματεύσει για την Τόχα. Αν κάποιοι λένε ότι η Τόχα είναι πλέον νεκρή και θα πρέπει να κοιτάξουμε νέα στοιχεία, e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο, θέματα προσαρμογή, το θέμα των ε, ε κερδοσκοπικών ε, τάσεων ε, για τι ισοτιμίε, θα προκληθεί εκ νέου διχασμός. Α προσπαθήσουμε με μερή τρόπο να χωρίσουμε και να εντάξουμε τον γύρο της Ντόχα και να αξιολογήσουμε θετικά τον γύρο της Ντόχα. Φυσικά χρειάζονται διευκρινήσεις, χρειάζονται στοιχεία ευελιξίας, σύμφωνοι, χρειαζόμαστε και διάφορες δυνατότητες διμερούς ή πολυμερούς ε, συνεργασίας, αλλά ότι αυτές οι εξελίξεις και αυτή η πρόοδος θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο είναι σαφές εν ώψη της μετανάστευσης και είναι σαφές ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, δεν είναι πάντα το ίδιο και οι χώρες ε, υποανάπτυξης έχουν ευθύνη και όλοι θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Λάρκιν. Uh, Συνάδελφοι, πιστεύω ότι το εμπόριο μειώνει την φτώχεια, δίνει δύναμη στι γυναίκε και δίνει και ευκαιρίε στου νέους μας. Ε, ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και οι πολίτε μα και οι καταναλωτέ μα θέλουν να φύγουν τα εμπόδια στο εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να κρύψω την απογοήτευσή μου λόγω την έλλειψη, της έλλειψης προόδου που έχει σημειωθεί σε επίπεδο ΠΟΕ και εν ώψη της 10 Υπουργικής Συνάντησης τον επόμενο μήνα και φαίνεται ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να γίνει καν μια κοινή δήλωση από πλευρά των μερών στον Αερόμπι. Είναι σαφές ότι η ατζέντα του, της Δόχα έχει αποτύχει, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε με κάποιο τρόπο την πολυμερή αυτή η ατζέντα και όλα τα σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια πολύ βασικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τι διεθνεί συμβάσει εμπορίου. Είναι σημαντικό όμως να αναγνωρίσουμε και τις άλλες φιλοδοξίε που είχε η Ντόχα. Προσπάθεια, για παράδειγμα, να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση για τι ε, πιο ε, αδύναμε χώρε στην ε, παγκόσμια αγορά και θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στους τομείς όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε αλλά φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα μπει στο πλαίσιο μιας διαφορετικής συμφωνίας πλέον. Άρα χρειάζεται μια νέα ατζέντα στα πλαίσια του ΠΟΕ που δεν θα συνδέεται με τις αποτυχίες του παρελθόντος και η οποία θα ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω προκειμένου να εξετάσουμε τον ΠΟΕ ως μια οργάνωση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του. Ωστότε τα μέρη θα αναγκάζονται να συνεργάζονται σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο για να υπάρχει ανάπτυξη και θέσει εργασία σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή που μπορεί να ασκήσει προκειμένου να προωθήσει αυτή την πολυμερή ατζέντα για να πετύχουμε επιτυχία για όλους. Έχετε μία μπλε κάρτα, κυρία Μακλάρκιν, από τον κύριο Κάρβερ. Να αποδέχεστε. Παρακαλώ κύριε Κάρβερ. Υπήρξε και ένα δεύτερο αίτημα, αλλά Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση δεν αποτελεί ένα παράδειγμα του πόσο μικρή είναι η επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου σε εμπορικές διαπραγματεύσεις και αυτό το θέτω και προς την κυρία Μάλμστρομ και αυτό δεν υποδεικνύει πόσο μεγαλύτερη επιρροή θα είχαμε αν βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δημοψήφισμα. Τα δευτερόλεπτα για να απαντήσετε σε αυτή την πρωτότυπη ερώτηση, κυρία Μακλάρκιν. The British people will decide whether they believe... Κοιτάξτε, οι Βρετανοί θα αποφασίσουν σύντομα αν θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπήρχε αυτή η απόφαση θα μπορούσαμε να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μόνοι μας. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε εμπορικές συμφωνίες για όλους και να υπάρχει, για να υπάρχει επιτυχία για όλους θα πρέπει να γίνει αυτό σε επίπεδο ΠΟΕ, ε, αναγκαστικά. Για την ομάδα φιλελευθέρων και δημοκρατών το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Στάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπέ. Όντως, η δέκατη υπουργική διάσκεψη που θα διοργανωθεί το Δεκέμβριο έχει ιδιαίτερη σημασία για μας και θα μας ε, δείξει πως η ατζέντα της ΔΟΧΑ, του αναπτυξιακή γυρίου της ΔΟΧΑ, θα προχωρήσει και κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Είμαστε τεθειμένοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και στο μέλλον. για τον αναπτυξιακό γύρο της Τόχα. Αλλά είμαι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε μια καινούρια βάση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει η παλαιά βάση που δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Θέλουμε μεγαλύτερη δέσμευση. Δεν ε, ήταν αυτό ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ενεργά υποστηρίξαμε τον αναπτυξιακό γύρο της ΔΟΧΑ Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε και την υποστήριξη άλλων από πλευρά διεθνού εμπορίου δε, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ε, παγκόσμιοι κανόνες για το εμπόριο. Αυτό θα δώσει βεβαιότητα, ασφάλεια, όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή κατακαιρματισμό. Οι λύσει του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα είναι πάρα πολύ σημαντικέ, θεωρούμε. Και αυτό γιατί συζητάμε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ακόμα και αν δεν καταλήξουμε σε μία λύση, θα συνεχίσουν οι συζητήσεις, οι και σε διμερές επίπεδο ή σε πολυμερές επίπεδο. Είναι σημαντικό, δε, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Να συζητήσουμε θέματα ουσίας. Αριστεράς, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Σόλτς. Κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μαχνίκ πριν από τα Χριστούγεννα θα μεταβεί στην Αφρική, στην Υπουργική Διάσκεψη, στο Νερόμπι και είναι ήδη σαφές ότι αυτό κατ' ουσίαν θα σημαίνει όδινεν όρος και έτε και μην. Αυτό δεν θα συμβάλλει σε τίποτα. Όποιος πραγματικά θέλει να πάει στο Ναϊρόμπι για ε, να επιτύχει κάτι, δεν θα καταφέρει τίποτα, θα σπαθήσει απλώς το χρόνο του. Γιατί τα 16 εκατομμύρια ε, δεν θα έπρεπε να ληφθούν περισσότερο υπόψη, αλλά εκείνο που ισχύει είναι ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανένα ότι τουλάχιστον αυτή η μία χώρα που θεωρεί τη δική τη διατροφή, τη διατροφή των πολιτών τη ε, σημαντικότερη από την ΠΟΕ, απορρίπτει όλα τα άλλα. Όχι, ο κύριος Λαμή απαιτεί ο ΠΟΕ επιτέλους ε, τη δουλειά της να την ε, προσφέρει ε, στους πολίτες, να την εντάξει στην κοινωνία των πολιτών. Με την, το γύρο της ΔΟΑ θα πρέπει να ξεπεραστεί η φτώχεια. Το γεγονός ότι ο στόχος αυτός ξεχάστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αυτό μας το επενθύμησαν τα πρόσφατα γεγονότα. Στο Ναερόμπι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή πορεία όσον αφορά τους στόχους και τους μηχανισμούς, την εμπορική πολιτική, τους κανόνες αυτό ακριβώς ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο γιατί πρόκειται για το μέλλον του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και ναι τελικά πρόκειται για τις προοπτικές ε, που έχουν ανοίξει με την ΤΟΧ. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για 2,5 λεφτά ο κύριος Μπούχνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε υπέρ του δικαίου εμπορίου. Αντίθετα με το δίκαιο εμπόριο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ε, δίκαιο παγκόσμιο φόρουμ όπου και οι αδύναμοι και οι δυνατοί θα μπορούν να κάσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν από κοινού λύσεις. Λύσεις που θα έχουν κάποιο όφελος για όλους τους εμπορικούς εταίρους. Εμείς, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ισχυρός εμπορικός εταίρος με μεγάλη επιρροή, ανδιαφυσβήτητα. Δεν πιστεύουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο είναι κάτι που θα πρέπει να καταπιέζει τους ε, ε, πιο αδύναμους ε, εταιρικούς εταιρούς μας. Και δεν είμαστε οι μόνοι. Ο ΠΟΕ προς τον σκοπό αυτό έχει προτείνει διαφορετική και διαφοροποιημένη προσέγγιση όλων των αναπτυσσόμενων χωρών. Βελτιωμένες συνθήκες πρόσβασης, για παράδειγμα, και σε ό,τι αφορά την αύξηση, για παράδειγμα, των εξαγωγών και εισαγωγών. Αλλά εσείς ζητάτε να γίνει κατανομή και διαχωρισμός των αναπτυσσόμενων χωρών σε κατηγορίες και οι χώρες οι οποίες ε, έχουν βελτιώσει τις ε, συνθήκες της οικονομίας τους τα τελευταία χρόνια να ανοίξουν πιο πολύ την αγορά τους. Αυτός ο διαχωρισμός ε, που θα ευνοούσε τους πιο ισχυρούς είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Το ψήφισμα λοιπόν επιβεβαιώνει την προσέγγιση του, της πολυμέρειας αλλά παράλληλα υποστηρίζει και πολυμερείς συμφωνίες όπως η ΤΙΖΑ οι οποίες υποσκάπτουν τον ΠΟΕ και δεν συμπληρώνουν όπως διατείνονται κάποιοι την ατζέντα του ΠΟΕ με διατάξεις για την πρόσβαση στην αγορά Με τον τρόπο αυτό λοιπόν στερούμε το οποιοδήποτε κίνητρο από τις πλούσιες χώρες να συνάψουν μια συμφωνία στο γύρο του Ντόχα. Το Ντόχα, η Ντόχα δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο ή θα το δεχτούμε ή θα το απορρίψουμε και θα το καταδικάσουμε. Και απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ξανασκεφτεί λοιπόν αυτό. Κάναμε κάποιες ε, τροπολογίες προκειμένου να είναι πιο δίκαιο και πιο αντικειμενικό το ψήφισμά μας. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η προσέγγιση να υποστηριχθεί. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Έθεριτς. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Έθεριτς. Τη δέχεστε. Κύριε Έθεριτς, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Thank you, thank you for accepting the blue card. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την κάρτα. Παρατήρησα ότι μιλήσατε για τους πιο αδύναμους εμπορικούς εταίρους δεν δέχεστε ότι οι αδύναμες χώρες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση διότι υπάρχουν φορολογικοί έλεγχοι μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων εμπορικών μπλοκ. Αν είχαμε ένα πιο δίκαιο σύστημα θα μπορούσαμε να έχουμε εμπόριο με τις χώρες αυτές και όχι ενισχύσεις. Ε, Στέκει όντως ότι τα γεωργικά μας προϊόντα μπορούμε να τα προσφέρουμε υπό όρους οι οποίοι δεν είναι αυτονόητοι για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή, πολλές από τις πολυμερείς συμφωνίες ουσιαστικά διαβρώνουν τις εθνικές αυτές γεωργικές οικονομίες. Άρα συμφωνώ σε αυτό και μόνο όμως, όχι με τα υπόλοιπα. Για την ομάδα ελευθερίας και άμεσης δημοκρατίας το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Earl of Mr. President. to get one thing in perspective... Θα ήθελα να σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε ως προστατευτικό μέσο ε, προστατευτικό οικοδόμημα και παραμένει τέτοιο. Πάντα θα είναι ένα τέτοιο ε, οικοδόμημα. Με ή χωρίς Ντόχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κόλλημα στο ελεύθερο εμπόριο. Και να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο θίξατε. Στον ε, τομέα της διατροφής, ο προστατευτισμός της Ευρώπης ε, πλήττει τον αναπτυσσόμενο κόμμα. Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι κλειστές ε, ως προς τη, τα αγροτικά προϊόντα λίγος πολύ. Επίσης, στην ουσία την ΚΑΠ την βάζετε πιο κάτω από την παραγωγή και αυτό μέσα στα πλαίσια και των επιδοτήσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων. Γι' αυτό και οι αγρότες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν μεγάλο πρωτογενή τομέα, πλήττονται και οι άνθρωποι που πλήττονται είναι οι πλέον ε, ενδέει στον κόσμο. Αυτό δεν είναι δίκαιο εμπόριο. Υπάρχουν και άλλες ε, συνέπειες. Ο προστατευτισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττει τους καταναλωτές στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτές εδώ θα πρέπει να πληρώσουν το υψηλότερο τίμημα για τρόφιμα και άλλα αγαθά. Ο καθηγητής Πάτρεκ Μίνφερτ του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ έκρινε ότι αυτό είναι το 8% ε, με βάση το κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, αν ε, προωθηθεί το Brexit, τότε το κόστος αυτό θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 8%. Ε, και πιστεύω ότι και σε άλλες χώρες θα είναι κάτι παρόμοιο. Άρα Πιστεύω ότι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν κάτι το θετικό για ολόκληρο τον κόσμο και ίσως αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για την ατζέντα της Ντόχα. Κύριε Έρλοτ Οφντάρμουθ, έχετε δύο μπλε κάρτες. Τρεις. Ήρθε και μια τρίτη τώρα στο τέλος. Θα δεχθώ όμως μόνο την πρώτη αν τη δέχεστε κι εσείς. Από τον κύριο Φιέλνερ. Τη δέχεστε? Okay. Κύριε Φιέλνερ, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να δίνω περισσότερες από μια μπλε κάρτα αναομιλητή. Ευχαριστώ. Εάν είσαστε τόσο αφελείς, κύριε Ντάρτμουθ, και θεωρείτε ότι όλες οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκλείψουν εάν ε, εξαλειφθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το ισόποσο όλων των κρατών μελών θα έφτανε σε υψηλότερους φόρους από τις δύο ε, ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την Ελβετία και την Ορβηγία, που έχουν πολύ υψηλότερες επιδοτήσεις. Παρακαλώ για την απάντησή σας. Υπάρχουν πολλέ χώρε που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Ελβετία και η Νορβηγία. Mm. Το γεγονό όμω είναι ότι αν υπάρχουν επιδοτήσει και ιδιαίτερα αγροτικέ, προσδιορίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Και αν ορίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, τότε, το, τότε θα εισακουστεί και ο καταναλωτής. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Φουντούλης. Μία εγγεγραμμένο κύριε πρόεδρε συζητάμε σήμερα για τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου και το πώς αυτός σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόμοιους οργανισμούς θα μπορέσει να σώσει τον κόσμο από τη φτώχεια μόνο που ε, για εμάς όλοι αυτοί οι οργανισμοί είναι μέρος του προβλήματος και μάλιστα μία από τις κύριες αιτίες του και προφανώς δεν είναι μέρος της λύσης. υπέρμαχοι ενός οικονομικού και κοινωνικού φιλελευθερισμού επιθυμείται οι παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις να καθορίζονται μέσα από υπερεθνικούς οργανισμούς με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση των κρατών οι κυβερνήσεις είναι οι μόνες που έστω και σε μικρό βαθμό ελέγχονται κάπως από τους πολίτες. αντίθετα οι υπερεθνικοί αυτοί οργανισμοί μεταβιβάζουν απλώς την εξουσία στις πολυεθνικές και στο μεγάλο κεφάλαιο ενώ προσποιούνται πως μοιάζονται και προσπαθούν να προστατεύσουν τους λαούς. στην πραγματικότητα οι οργανισμοί αυτοί είναι που προωθούν την απελευθέρωση των αγορών από κάθε είδους εμπόδιο και έλεγχο με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και για ολόκληρε κοινωνίες επιπλέον οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταραίουν αδύναμες να αντιπαρατεθούν στην επέλαση των μεγάλων ομίλων που υποστηρίζονται ενεργά από τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου την ίδια στιγμή μάλιστα που όλοι προσποιούνται πως ενδιαφέρονται για αυτές μην μπορώντα όμω να κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο δεν αρκεί στον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου να ελέγξει την οικονομική δραστηριότητα όλων των κρατών. επιδιώκει να επιβάλλει τι απόψει του σε κάθε πτυχή τη κοινωνία στη διαχείριση τη δημόσια διοίκηση στη φορολογική πολιτική στην εκπαίδευση στι κοινωνικέ πολιτικέ και σε θεσμικέ μεταρρυθμίσει. ε λοιπόν όχι! καμία διευκόλυνση για το διεθνές τοκογλυφικό κεφάλαιο καμία παραχώρηση σε όσους καταστρέφουν έθνη και λαού για το χρήμα. για εμάς του έλληνες εθνικιστές η μόνη θετική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου θα ήταν να αυτοδιαλυθεί. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για την καλή πρόταση ψηφίσματος. Η απελευθέρωση του εμπορίου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε την ε, διεθνή ανάπτυξη. Και το διεθνές εμπόριο λοιπόν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο εργαλείο για τις ε, λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Η σημασία δε του εμπορίου για την βιώσιμη ανάπτυξη έχει ε, αναγνωριστεί και στην ατζέντα του 2030 και έχει αναγνωριστεί ένα, ένα σημαντικό εργαλείο για την ε, συνολική ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Και είναι συμβολικό λοιπόν το γεγονό ότι η δέκατη Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα τόνισε τη σημασία της πολυμέρειας καθώς και των ε, προσωρινών λύσεων όπως είναι οι περιφερειακές και πολυμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες. Ωστόσο, προκειμένου να πετύχουμε κάποια στο θετικά αποτελέσματα στην υπουργική αυτή διάσκεψη, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των ταχαίως ε, αναπτυσσόμενων χωρών μεσαίων εισοδημάτων και θα πρέπει λοιπόν να γίνουν περαιτέρω βήματα για την απελευθέρωση του εμπορία και για την επιτεύξη των βιώσιμων στόχων από την ατζέντα του 2030. Θα, δώσουμε επίσης, θα πρέπει να δώσουμε σημασία για την μεταρρύθμιση της αρρώγης του εμπόριου, για την διευκόλυνση του εμπορίου, για να βοηθηθούν οι χώρες να αυξήσουν το δυναμικό τους ως προς το εμπόριο και έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το, το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 68 δις αναέτος και αυτό θα ωφελούσε κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω την ε, επικύρωση της συμφωνίας αυτής προκειμένου να τεθεί σε ισχύ πριν από την τακατυπουργική. Δύο αιτήματα για μπλε κάρτα. Το πρώτο είναι από τον κύριο Ρούμπικ. Επαναλαμβάνω ότι θα δέχομαι μόνο ένα αίτημα αναομιλητή, ένα μπλε κάρτα. Επομένω, το αίτημα τη κυρία Γκραπίνη ήρθε δεύτερο την επόμενη φορά. Ε, δέχεστε την ε, μπλε κάρτα του κύριου Ρούμπικ. Κύριε Ρούμπικ, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφό μου τον κύριο Στήρ το εξή το γεγονός ότι οι εμπορικές διευκολύνσεις επιφέρουν μεγαλύτερη ευημερία στις ανεψόμενες χώρες, αυτό είναι σαφές. Αλλά το πρόγραμμα Aid for Trade είναι πολύ σημαντικό, κυρίως να εστιάζεται στις χώρες εκείνες από τις οποίες προέρχονται οι προσφυγικές ροές. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτή η συζήτηση τώρα στην Κένια και δεν πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι τους ανθρώπους εκείνους έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν στις πατρίδες τους. Δευτερόλεπτα Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, ασφαλώς συμφωνώ μαζί σας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι ενδεχομένω να ισχύει έμεσα, αλλά στο ψήφισμα αυτό τονίζεται εξίσου. Και γι' αυτό λοιπόν δήλωσα ότι θα πρέπει να δώσουμε σημασία στη Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, προκειμένου να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν το εμπορικό δυναμικό και να καταπολεμήσουν την φτωχία, προκειμένου να, τη προκειμένου να μπορούν να ε, θρέψουν τον κόσμο τους. Για ένα λεπτό η κυρία Ροντρίγκεθ Πινιέρο. Ευχαριστώ. Δέχομαι την εξαιρετική εργασία των δύο εισηγητών. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να επιδίδεται στις, ε, στην πρόθεση των πολυμερών σχέσεων μέσα στα πλαίσια των εταίρων του ΠΟΕ. Δεν ε, πρέπει να οροβούμε. Θα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση έγκριση της Συμφωνίας Διευκολύσεων και να ζητήσουμε να ε, προωθήσουμε ένα πολύ, μια πολύ ανοιχτή ε, ατζέντα της Ντόχα με έναν οδικό χάρτη στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθούν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού, ιδιαίτερα προς τα αγροτικά προϊόντα και τις επιδοτήσεις. Οι αναδιόμενες οικονομίες να έχουν τη δική τους, το δικό τους ποσοστό ευθύνης μέσα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου και χρειάζεται και μεγαλύτερη ευελιξία των προηγμένων χωρών. Θα πρέπει βεβαίως να μεταρρυθμιστεί και ο ΠΟΕ, έτσι ώστε να αυξηθεί ο ρόλος της διακυβέρνησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Χένκελ. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως ε, θα ήταν ε, πάρα πολύ ωραίο το να έχουμε τέτοιου είδους ε, γύρους του ΠΟΕ που ε, να μην τσακωνόμαστε πλέον για το TTIP και για οτιδήποτε άλλο. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω κάτι άλλο. Κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχει παγκοσμιοποίηση και γιατί είναι τόσο σημαντικό το ελεύθερο εμπόριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν αφορά μόνο τα εμπορεύματα, τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, αλλά και τις ιδέες και τις αξίες και το οφείλουμε στην παγκοσμιοποίηση το γεγονός ότι σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζονται ως ένα οικουμενικό θέμα, μια οικουμενική ευκαιρία. Βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει και πολύ περισσότερη δημοκρατία στον κόσμο από ότι οποτεδήποτε κατά το παρελθόν. Και αυτό το οφείλουμε στην παγκοσμιοποίηση. Άρα δηλαδή θα πρέπει να στηρίξουμε τον ΠΟΕ και το εμπόριο γιατί το εμπόριο οδηγεί σε μεγαλύτερη ευημερία. Και κατά τα άλλα ε, κυρίες και κύριοι θεωρώ ότι ότι το ευρώ οδηγεί μόνο σε τσακωμούς στην Ευρώπη, διαφωνείς, γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί το ευρώ. Έχω δύο αιτήματα για μπλε κάρτα. Το πρώτο από τον κύριο Earl of Dartmouth και το δεύτερο από τον κύριο Σάνι. Αλλά λέω κύριε Earl of Dartmouth ότι εσείς ήδη μιλήσατε, μη βιάζεστε, εσείς ήδη μιλήσατε, απαντήσατε και σε μια μπλε κάρτα, επομένως θεωρώ δικαιότερο να δώσω το δικαίωμα για μπλε κάρτα αυτή τη φορά στον κύριο Σάνι. Κύριε Χένκελ, δέχεστε την, το αίτημα για μπλε κάρτα του κύριου Σάνι. Παρακαλώ κύριε Σάνι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η δική μου ερώτηση προς τον συνάδελφο είναι η εξής. Αν θεωρητικά όλες αυτές οι διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες περάσουν. Πιστεύετε ότι μπορούν αυτές οι περιφερειακές συμφωνίες να καταστούν μια παγκόσμια συμφωνία. Δεν το πιστεύω, αλλά θα ήθελα να ακούσω τι πιστεύετε. Απαντήστε κύριε Κοιτάξτε, συμφωνώ και εγώ πιστεύω ότι αν ε, είχαμε μια ιδανική παγκόσμια συμφωνία δεν θα χρειαζόμασταν αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Πρέπει όμως να πούμε ότι ο αριθμό ε, όλων των διμερών συμφωνιών στο σύνολό τους συνέβαλαν περισσότερο από ότι ο ΠΟΕ. Παρ' όλα αυτά για μένα ο στόχος παραμένει σαφής. Ο ΠΟΕ πρέπει να στεφτεί από επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και στην περίπτωση αυτή δεν θα χρειαζόμαστε πλέον αυτές όλες τις άλλες συμφωνίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπέ, κύριε Επιτροπέ. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν κόσμο που όλε οι πόρτε θα είναι ανοιχτέ για τι επιχειρήσει μα και το παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο αποτελεί το κλειδί για τι πόρτε αυτέ. Αν θέλουμε να είναι ισχυρή η Ευρώπη, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ε, αφαίρεση όλων των ε, φραγμών και στα πλαίσια του ΠΟΕ και εκτό του ΠΟΕ. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να μπει μία γραμμή κάτω από τα τελευταία 14 χρόνια των συζητήσεων στα πλαίσια του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα και να προχωρήσουμε προς τα μπροστά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία νέα στρατηγική για την Ντόχα και για τον θεσμό της Δόχα. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν στην παρούσα φάση για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Καταρχάς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο γύρος αυτός σε ένα κάποιο φόρουμ προκειμένου να συνεχιστεί και να εξελιχθεί η πολυμερής ατζέντα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ηγείται τη συζήτηση αυτή. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση όλων των μελών προκειμένου να υπάρχουν κάποια πραγματικά αποτελέσματα από τις συνομιλίες αυτές ακόμα και αν αυτά τα αποτελέσματα είναι πιο μικρά από αυτά που αρχικά ελπίζαμε. Κατά δεύτερον, στη συνέχεια, προκειμένου να υπάρξει μια πολυμερής ατζέντα. Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουμε στα πλαίσια της πολυμερούς ατζέντα για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και η διάσκεψη στον Αερόμπι θα πρέπει να έχει ως στόχο το να αποδεχτούμε ρεαλιστικά αποτελέσματα στα πλαίσια της Ντόχα αφενός, αλλά και να τεθεί και ένας φιλόδοξος τρόπος για τα πλαίσια του ε, γενικότερα. Έχετε μια μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπίνη. Τη δέχεστε? Ε, δέχεστε τα συγχαρητήρια του συναδέλφου σας, αλλά ακούστε με και μένα, δέχεστε την μπλε κάρτα. Παρακαλώ κυρία Γραπίνη, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Συμφωνώ με τους εισηγητές, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, συνάδελφε, κατά πόσο νομίζετε ότι ο ΠΟΕ θα πρέπει να έχει διαφορετική εμπορική ατζέντα έτσι ώστε οι δυνατές χώρες μπαίνοντα στον ΠΟΕ να μην φτάσουν σε αθέμητο ανταγωνισμό που ζούμε πολλές φορές από πλευρά της Κίνας η οποία βάζει στο εμπόριο μη ελεγχόμενα προϊόντα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος για την προστασία του καταναλωτή. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. Έχετε 30 δεύτερα για την απάντηση. Thank και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρόκειται πραγματικά ένα ορόσι, για ένα ορόσημο όπου θα πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Είναι ένα θέμα κρίσιμης σημασίας η προώθηση της ατζέντα αυτής. Δεν έχει νόημα να έχουμε μόνο δίμερις ή περιφερειακές ε, συναντήσεις και συμφωνίες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Σάντσες Ντέι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο γύρος της Ντόχα αντιμετωπίζει μεγάλες ε, προκλήσεις. Δεν είναι απλό γιατί έχουμε ως αντιπαραβολή τις πλούσιες με τις φτωχές χώρες. Είναι δύσκολο να φτάσουμε σε συνενέσεις από τις οποίες θα ευεργετηθούν όλοι, ιδιαίτερα οι κάτοικοι του Νότου. Αυτό το βλέπουμε και με το ΤΠΠ και με το ΤΤΙΠ. Βλέπουμε ότι ζούμε την ηγεμονία των πλουσίων. Θα πρέπει στην Αϊρόμπη να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να φτάσουμε σε ένα σωστό εμπορικό πλαίσιο όπου να εκπροσωπούνται όλοι το διεθνές εμπόριο θα πρέπει να βοηθήσει για να καταπολεμηθεί η φτώχεια και οι κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον. Αυτό το νόημα έχουν αυτές οι μακροδιαπραγματεύσεις. Λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μπεγκίν. Grazie, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην συνάντηση στο Εναρόμπι τίθεται σε συζήτηση το ίδιο το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστημα το οποίο η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε σκοτώνουν λόγω του TTIP, του TISA και άλλων συμφωνιών. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, υπάρχει ο πολυμερισμός ε, ως λύση, αλλά το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί γιατί πρέπει να το μεταμορφώσουμε. Ε, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις πιο φτωχές χώρες, να τις βοηθήσουμε συνεχίσουμε, αλλά θα πρέπει επίσης ε, να ξεχάσουμε αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα σε χώρες σε ανάπτυξη και αναπτυγμένες. Η Κίνα και η Ινδία μπορούν να στείλουν κάποιον στο φεγγάρι, αλλά θεωρούνται αναπτυσσόμενες χώρες και κατόπιν τούτου υποφελούνται. Πρέπει να ε, βοηθήσουμε τους ε, πιο φτωχούς. Ήδη προσφέρουμε αρκετά, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον ΠΟ για να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία για τους κανόνες προέλευσης. Βεβαίως αυτά μπορεί να λυθούν καλύτερα σε πολυμερές επίπεδο. Πρέπει να προσπαθήσουμε στο Ναϊρόμπι να έχουμε επιτυχία για να μην ακολουθηθεί η μοίρη των συμφωνιών TTIP. Άρα δηλαδή στην περίπτωση αυτή αν δεν πετύχουμε θα έχουμε χάσει τα πάντα. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Φίσας Αϊσέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους ε, συναδέλφους ε, Λάγκια και Σάλπα για αυτή την εξαιρετική εισήγηση εν ώψη της Υπουργικής Διάσκεψης στην Κένια το Δεκέμβριο. Η δημιουργία του ΠΟΕ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς ένα ολοκληρωμένο εμπορικό σύστημα και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, με μεταβατικές οικονομίες μπορούν να προωθήσουν τη δική τους ανάπτυξη. Μέσω του ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι θέλει να ορίσει ένα διεθνές ε, εμπορικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια και των πολυμερών και περιφερειακών ε, συμφωνιών. Μιλάμε για ένα διεθνές εμπορικό σύστημα το οποίο συνεχώς αλλάζει. Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο σύστημα, με νέες χώρες και μια νέα πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να υποστηρίξουμε μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για να υπάρχει πιο σωστό και ανοιχτό εμπόριο και να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε η Επίτροπος και επεσήμεναν και οι άλλοι συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η συμβολικότητα του γεγονότος ότι είναι η πρώτη διάσκεψη που γίνεται στην Αφρική και θα πρέπει να είναι αυτό μια ευκαιρία, να δοθεί ως μια ευκαιρία για τον γύρο της Δόχα και να τονίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται αναπτυξιακά στοιχεία στη διάσκεψη αυτή, την Υπουργική. Καταρχά, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ηθική και διαφοροποιημένη προσέγγιση που αποτελεί ε, την, ε, τον πυρήνα κάποιων συζητήσεων στην Υπουργική Διάσκεψη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε για το άνοιγμα του εμπορίου. Και όπω είπαν και οι άλλοι σήμερα το απόγευμα, όλοι καλώ ορίζουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου και θα πρέπει αυτό να δοθεί ως μήνυμα πριν από την Υπουργική Διάσκεψη. Ξέρω ότι είναι έντονη η εργασία προς την κατεύθυνση αυτής. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ουσιώδου σημασία πριν το ένα αερόμπι. Και επίσης, ο κύριος Ρούμπι, αν δεν κάνω έθεσε το θέμα του να γίνουν δεσμεύσεις από πλευρά των κρατών μελών για το Aid for Trade. Και κάποια κρατημέλη πριν από κάποια χρόνια ε, ουσιαστικά γνώρισαν αυτές τις εκκλήσεις. Τέλος, αν και αυτό δεν αποτελεί θέμα της Υπουργική Διάσκεψης, θα ήθελα να ευχαριστήσω επ' ευκαιρίας ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση του Συμβουλίου του ΠΟΕ για τη θέση των λιγότερων αναπτυγμένων ε, χωρών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση για τα φάρμακα. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Βαουένσα. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό είναι πολύ επίκαιρο για να δείξει την πρόθεση της ατζέντα της Δόχα για όφελος όλων Υποστηρίζεται λοιπόν οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ και αυτή η μεταρρύθμιση ελπίζουμε ότι θα πετύχει ένα πιο ανοιχτό, πιο διαφανές ε, εμπορικό σύστημα, με λιγότερες ε, ε, διακριτικές μεταχειρήσεις διαφόρων χωρών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα του ΠΟΗ για να προσαρμοστεί στα πραγματικά προβλήματα, στην πραγματικότητα, να είναι πιο ρεαλιστικό και να εκπληρώσει τον ρόλο του για την βοήθεια των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων και επίσης των καινοτόμων startups, νέων εταιριών, νέων επιχειρήσεων. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξει και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις χώρες που ανάπτυξη. Υποστηρίζει τους σωστούς ορισμούς για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος και για τις αναδυόμενες οικονομίες. Και αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος, για παράδειγμα, της Κίνας στο θέμα του ΠΟΕ. Και τέλος πιστεύω ότι οι διατάξεις του ψηφίσματος έχουν ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την απελευθέρωση των σχετικών πολιτικών. Τούτων λεχθέντων λοιπόν υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό απόλυτα και πιστεύω ότι θα είναι επωφελές για όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επόμενη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα θέματα της πολυμέρειας, ε, για τον ΠΟΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών. Η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνάψει σημαντικές συμφωνίες που ακόμα είναι σε φάση διαπραγμάτευσης. Το βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής ε, είναι να δοθεί όθηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα πολυμερών συμφωνιών που θα είναι και το οδηγό νήμα για την παγκοσμιοποίηση. Όσον αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατ' ουσίαν ε, θα θέσει τα χαρτιά της στο Νερόμπι. Αυτή η πρώτη συμφωνία προβλέπει μια καινοτόμα προσέγγιση όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό θα επιτρέψει να ε, επιλέξει κανείς και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Εύχομαι λοιπόν στο Ναϊρόμπι να υπάρξει μια αποτελεσματική στρατηγική που θα διευκολύνει το πολυμερές εμπόριο. έχει για δύο λεπτά ο κύριος Φιέλνερ. Eh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και εσάς κυρία Επίτροπε. Το ελεύθερο εμπόριο αποτελεί ε, το πιο σημαντικό εργαλείο για να, να πετύχουμε την ευημερία. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικές αυτές οι συμφωνίες εμπορίου, ελεύθερο εμπορίο. Αλλά ο γύρος της Δόχα μας έχει ταλαιπωρήσει τόσα πολλά χρόνια και πραγματικά δεν φαίνεται να σημειώνεται πρόοδος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ε, πρόοδο στο Ναϊρόμπι και για να σας πω τρεις λόγους γιατί είναι τόσο σημαντικό να υπάρξει εξέλιξη. Καταρχάς για να προχωρήσει το παγκόσμιο εμπόριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοιες επικίνδυνες εποχές. Κατά δεύτερον, τώρα χρειαζόμαστε πιο πολύ από ότι ποτέ παγκόσμιους ε, κανόνες για το εμπόριο, για τις τελωνιακούς δασμούς, προκειμένου να καταργηθούν τα εμπόδια που υπήρχαν ως σήμερα. Πραγματικά είναι δυσδιάκριτη πλέον η κατάσταση. Το εμπόριο δεν πρέπει να γίνεται πιο δύσκολο, πιο ακριβό, πιο περίπλοκο. Και κατά τρίτον, το θέμα αυτή τη στιγμή που διακυβεύεται είναι και η ίδια η αξιοπιστία του ΠΟΕ. Δεν πρέπει το θέμα να είναι μόνο η επίλυση των ε, διαφόρων διενέξεων. Θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και όπως είπε λοιπόν η Επίτροπος, δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα ολοκληρωθεί ο γύρο αυτό, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον οι τομεακέ συμφωνίε θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Είναι δυνατόν. Θα πρέπει εκεί να σημειωθεί πρόοδο. Για παράδειγμα, μια παγκόσμια συμφωνία για προϊόντα πιο φιλικά προ το περιβάλλον. Εκεί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει τα μάλα και ελπίζω ότι οι τελωνιακοί δασμοί για τέτοια προϊόντα μπορούν να καταργηθούν. Αυτό χρειάζεται πραγματικά. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Φερέιρα. Τη δέχεστε. Κύριε Φιέλνερ, έχετε μία μπλε κάρτα. You, you have a blue card from Mr. Ferreira. Do you, do you accept it? Okay. Κύριε Φερέιρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριος Φιέλνερ στη ουσία είναι υπέρ της φιλελευθεροποίησης της αγοράς. Ε, ισχύει κάτι τέτοιο γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή οι χώρες ΑΚΕ, ε, προσπάθησαν να αντισταθούν στις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Αν είναι τόσο καλές, γιατί αντιστάθηκαν οι χώρες αυτές και δεν τις δέχτηκαν δηλαδή να τους επιβάλλουν τέτοιες ε, πολιτικές οι βιομηχανικές χώρες, οι πολύ δυνατές χώρες. για την απάντηση. Thank you very much. If that was true... Σας ευχαριστώ. Αν αυτό δεν μπορεί να συμφωνούσα μαζί σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλές από τις χώρες αυτές είναι στο δρόμο προς μια συμφωνία τέτοια εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι γεγονός. Και βλέπουμε ότι σε τέτοιες ε, εποχές σήμερα έχουμε πιο λίγους φτωχούς ε, από άρα στον κόσμο. Και αυτό όχι χάρη στις κομμουνιστικές ιδέες, χάρη στο ελεύθερο εμπόριο και τίποτα άλλο. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές ε, διότι η έκθεση αυτή εκφράζει ρεαλιστικά το γεγονός ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία τελική όθεση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και για να φτάσουμε σε απτές λύσεις. Επειδή υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια για το πώς σκεφτόμαστε την παγκοσμιοποίηση, η οποία έχει και αρνητικές πλευρές, όπως ζούμε τις τελευταίες μέρες, το Ναϊρόμπι αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία διότι θα ήταν η θετική πλευρά της παγκοσμιοποίησης εκεί όπου ενισχύουμε το πολυμερές σύστημα μέσα στα πλαίσια δίκαιων συμφωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Μας ενδιαφέρει η οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η κοινωνική και η περιφαλλοντική και η, ανθρώπινη ανάπτυξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση στο Ναϊρόμπι και αυτή είναι και η προτεραιότητά μας όπως εκφράζεται στο ψήφισμα. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Βέντα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Επιτροπέ. Όπως αναφέρατε, η 10η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ θα λάβει χώρα για πρώτη φορά σε αφρικανική χώρα και η διακήρυξη της ΔΟΧΑ υπογραμμίζει με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ του εμπορίου και της ε, εξέλιξης. Και είναι ενδιαφέρον από πλευρά ε, των αναπτυσσόμενων χωρών το γεγονός ότι αυτό παραμένει θέμα διαπραγμάτευσης γιατί δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Η κατάργηση λοιπόν των εμπορικών αυτών εμποδίων και η καταπολέμηση δημιουργία τέτοιων καινούριων εμποδίων συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και η σε ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Τόχα μπορεί να έχει διαφορά μέχρι και 300 δισεκατομμύρια ΕΠΕ Το πιο μεγάλο τμήμα εξ αυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό λοιπόν θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της στόχιας στις χώρες αυτές. Στον γύρο αυτών των διαπραγματεύσεων, λοιπόν, οι πιο πολλές αναπτυγμένες ε, χώρες θα πρέπει να αναλάβουν πιο πολλές ευθύνες ό,τι αφορά τις δράσεις τους και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει υπεύθυνη αντιμετώπιση η οποία θα αποτυπώνει τις ανάγκες των πιο φτωχών χωρών. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν στο εμπόριο είναι κάτι το απαραίτητο, ιδιαίτερα στη θέμα και στον άξονα τους, της γεωργίας, των γεωργικών προϊόντων. Αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν αφαιρώντας τους ποσοτικούς ε, περιορισμούς και τους τελωνιακούς δασμούς. Και αυτό λοιπόν θα διευκολύνει τους απλούς ανθρώπους στην καθημερινή του ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είμαστε επιτυχείς. Ένα λεπτό, ο κύριος Σίλβα Περέιρα. Κύριε Πρόεδρε, η Επίτροπος Μάλμστρεπ μας είπε ότι έχουμε ένα μήνα μπροστά μας μέχρι την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ. Όμως οι προπαρασκευαστικές εργασίες δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές εν ώψη μιας επιτυχίας στο Ναϊρόμπι. Σε, γιατί καμία ατζέντα περιφερειακής ε, φύσης ή υφής δεν αντικαθιστά τις πολυμερείς σχέσεις. Εδώ μιλάμε για πολυμερείς σχέσεις και δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία εάν στην ε, προπαρασκευαστική φάση δεν ε, δημιουργήσουμε τις σωστές συμμαχίες για να υπάρχει πιο δίκαιο εμπόριο που να χρησιμοποιηθεί σωστά. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ναϊρόμπι έτσι ώστε να ε, δημιουργήσουμε αυτές τις σωστές συμμαχίες για να υπάρξει επιτυχία στη διάσκεψη. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εγγεγραμμένων ομιλητών και περνούμε στην διαδικασία του Catch the Έχω δεχθεί οκτώ αιτήματα για τη διαδικασία του Catch the Θα προχωρήσω με την γνωστή μέθοδο ένας ομιλητής, ο πρώτος αναπολιτική ομάδα. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή είναι επιγόντως απαραίτητη. Βρισκόμαστε την ψηφιακή εποχή και εξακολουθούμε να κάνουμε συζητήσεις ε, για το τι θα γίνει με, τη, με το γύρο της ΔΟΧΑ. Ο κόσμος ε, έχει αλλάξει ριζικά και όσον αφορά το Aid for Trade θα πρέπει να βοηθήσουμε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε τους ε, ανελεύθερους επαγγελματίες εκεί όπου επικρατεί η φτώχεια. αυτό θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος μας και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά για σε πάρα στη διοίκηση, στα τελωνία υπάρχουν εμπόδια για ελεύθερο εμπόριο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικός να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν και πάλι επαρκή τροφή. Ε, Πώ μπορούμε να δώσουμε αρκετά τρόφιμα στα 10 δις ανθρώπων που τα χρειάζονται. Ε, γι' αυτό λοιπόν Γεωργία και Aid for Aid αυτό είναι ένα πακέτο επιγόντως απαραίτητο. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Καπούτο. Grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέσα στα πλαίσια των παρασκευαστικών εργασιών της Ντόχα είναι μεγάλης σημασίας να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση μέσα στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών για να βοηθήσουμε τις πλέον αδύναμες χώρες για να μπορούν να ανταποκριθούν. Νομίζω ότι η γέφυρα που συνδέει τις δύο αυτές πραγματικότητες είναι πολύ ευάλωτη. Θα πρέπει λοιπόν ο γύρος της Ντόχα να αντιμετωπίσει τις ανισότητες του συστήματος μέσα στα πλαίσια της εποπτείας ε, της πολυμέρειας των ε, συμφωνιών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και διμερείς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το άρθρο 20 της Συμφωνίας του Μαρακές έτσι ώστε να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος, διατροφική ασφάλεια, ευζοία των ζώων έτσι ώστε να υπάρχει ένα βιώσιμο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών. σε ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η αναπτυξιακή ατζέντα της ντόχα οφείλει να αποσκοπεί στην οικονομική μεγέθυνση στη θέσπιση κανόνων για τη διευκόλυνση ενός δικαίου εμπορίου και στη μείωση των ανισομεριών στο διεθνές σύστημα εμπορικών συναλλαγών. ωστόσο αυτό που τελικά συμβαίνει στην πράξη είναι η πλήρης και ανεφόρον απελευθέρωση του εμπορίου που οδηγεί στην αποβιομηχάνηση στη μείωση της απασχόλησης και στις οικονομικές κρίσεις. παράλληλα ζημιωμένοι βγαίνουν και οι αγρότες ενώ επιπλέον ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου όχι μόνο χαρακτηρίζεται από βαθύ δημοκρατικό έλλειμμα αλλά απέτυχε να συμβάλει στην αποτροπή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. είναι επομένως αναγκαίο να διαμορφωθούν δίκαιοι και ισορροπημένοι εμπορικοί κανονισμοί που να υπηρετούν την κοινωνική δικαιοσύνη. επιπλέον θα πρέπει κάθε κράτος να διατηρεί την κυριαρχία του στη ρύθμιση των οικονομικών του σχέσεων καθώς και στην κατανομή των πόρων στους διάφορους δημόσιους τομείς για να μπει έτσι φραγμός στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων μέσω των ανισομερών εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice, svjetska trgovina mora postati instrument i το παγκόσμιο εμπόριο θα πρέπει να καταστεί ένα εργαλείο για την ανάπτυξη και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει για μας λοιπόν, θα πρέπει να θεωρήσουμε φυσικά καλύτερα να, να γίνει κάτι προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο αντί να δίδεται ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι καλύτερα να καταστούν οι οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών και οι αγρότες επιτυχείς προκειμένου να μην τους δίνουμε τα ψάρια αλλά να τους μάθουμε να ψαρεύουν οι ίδιοι. Δεν επαρκούν λοιπόν οι πόροι για να συνεχίσουμε παόριστο να τους βοηθάμε. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να μάθουν να είναι αυτάρχεις και θα πρέπει λοιπόν με τον τρόπο αυτό να αναπτυχθεί το παγκόσμιο εμπόριο και εμείς μπορούμε έτσι να αναπτυχθούμε γιατί δάλος, δεν θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριοι βουλευτές, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η επιτυχία του Μπαλί ε, ήταν κατά των φτωχών. Δυστυχώς ε, τα πλήρωσε όλα η αγροτιά, γιατί παρά τα όσα είπατε πολύ, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όσο πιο ελεύθερο είναι το εμπόριο, τότε ο πλούτος συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια. Στο Κανκούν το 2013 ο κύριος Λίκιου Χάι, ένας αγρότης, ζήτησε από τον ΠΟΕ μία πιο αξιοπρεπή ζωή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ήρθε καιρός να θέσουμε τέλος στον ΠΟΕ. Μιλήσατε κι εσείς για την ΚΑΠ η οποία στην ουσία καταστρέφει χιλιάδες εκατομμύρια αγρότες και δείχνει ότι ο ΠΟΕ είναι μεγάλη αποτυχία για όλο τον κόσμο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch Το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής έχει η κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ επίσης και τους συζητητές για όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Ακόμα και αν υπάρχουν κάπου διαφωνίες, ε, υπάρχει από ό,τι φαίνεται υποστήριξη για την πρόταση ψηφίσματος. Η Κομισιόν και εγώ προσωπικά είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το πολυμερές σύστημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε ζωντάνια στον ΠΟ, γιατί πράγματι χρειαζόμαστε ένα διεθνές φόρουμ όπου θα ισχύουν διεθνείς κανόνες ε, και εκεί θα συμμετέχουν όλα τα κράτη, όλα τα κράτη του κόσμου. Τώρα έχουμε 161. Είναι απαραίτητο να γίνουν συζητήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και χρειάζεται για αυτόν τον λόγο και ενέργεια. Αλλά βεβαίω πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στον Ναϊρόμπι. Γίνεται λόγο για την Doha Development Round. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ανάπτυξη. Και πράγματι κύριε Περέιρα έχουμε συνεργαστεί στενά ε, και με άλλε χώρε, με τι χώρε ΑΚΕ για να μπορέσει μπορέσουμε να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε το θεματολόγιο μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πιο φτωχές χώρες του κόσμου θα επωφεληθούν από αυτή τη συμφωνία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αναζητάμε να βρούμε λύσεις στον ανταγωνισμό των εξαγωγών. Ε, οι εξαγωγές και η στρέβλωση των ισχύσεων αυτό βλάπτει τις φτωχές χώρες. Βεβαίω αυτό που ψάχνουμε επίσης είναι να δούμε λιγάκι τους κανόνες προέλευση, ε, και αυτό που ψάχνουμε επίσης είναι να υπάρχει και διαφάνεια στο σύστημα. Ε, βεβαίως αυτό δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ και διαφορετικές φωνές. Δουλεύουμε λοιπόν πολύ σκληρά στη Γενέβη, όπως σας είπα, και θα ήθελα να πω στους ε, συναντέλφους από το και που φύγαν όμως όλοι, δεν υπάρχει κανείς εδώ από αυτούς πια, ότι ε, θα πρέπει ε, να μιλάμε με μία φωνή όπως συμβαίνει στον ΠΟΕ. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχουν 161 χώρες. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές απόψεις για το κατά πόσο να έχουμε μεταρρυθμίσει την κοινή αγροτική πολιτική όχι. Αλλά αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εισαγωγέ τροφίμων από τι φτωχέ χώρε και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τι ενισχύσει εξαγωγών. Γι' αυτό λοιπόν και πιέζουμε να υπάρξουν καταργήσει στο Ναϊρόμπι, ε, στη Βραζιλία και αλλού. Επίση ε, θα δουλέψουμε σκληρά για άλλε τρει εβδομάδε. Ε, το αποτέλεσμα ακόμα δεν είναι σαφέ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι την τελευταία στιγμή στο Ναϊρόμπι για να επιτύχουμε συμφωνία. Ναι κύριε Φέλνερ, Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και τις ε, διευκολύνσεις εμπορίου ε, και τα πράσινα εμπορεύματα. Ε, έχουμε κάνει κάποια πρόοδο στην Τίζα. Θα δούμε τι θα γίνει στο Ναερόμπι και προσβλέπουμε στο να ε, συναντηθούμε με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι παρόν ε, στο Ναερόμπι. Μετά τα Χριστούγεννα ε, θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε, να δούμε τι θα έχει γίνει με τα συμπεράσματα. Και εν πάση τόση, αν κάτι αποτύχει, αυτό δεν θα οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 5η 26 Νοεμβρίου του 2015. Good evening, colleagues. Uh,